organization. Good afternoon everybody. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σε αυτή την ε, διάσκεψη ψηλού επίπεδου για τη διαχείριση της μετανάστευσης που διοργανώνει το Ευρωκοινοβούλιο μια μέρα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το θέμα αυτό έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα μπορείτε να μιλήσετε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Υπάρχει διερμηνία. Και εγώ θα μιλήσω τη δική μου μητρική γλώσσα, την Ιταλική σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο πολύ ε, στην ε, αίθουσα αυτή, στη, για την αθρώα αυτή προσέλευση. Η ημερομηνία και ο τόπος της εκδήλωσης δεν είναι τυχαίοι. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τους πρόσφυγες. Αύριο ξεκινά ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα μπορούσε επιτέλους να σημάνει μία καμπή στην πολιτική μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή της θητείας μου Δήλωσα ότι θα αφιερώσω τα δυόμιση ε, αυτά χρόνια προεδρία στο Κοινοβούλιο για να γεφυρώσουμε τα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για να γίνει αυτό πρέπει να ακουστεί ισχυρή και στεντόρια η φωνή του Κοινοβουλίου όπου ε, έχουν την έδρα τους 751 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Σήμερα στην Ολομέλεια βρίσκονται μαζί μας όχι μόνο οι εκπρόσωποι των θεσμών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Αφρικής, ε, ταυτόχρονα επίσης και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και διεθνείς οργανισμούς και τόσοι άλλοι φορείς που προσπαθούν να βρουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα τοπικές ε, αρχές, αρχές τοπικής αυτοδίκησης, δήμαρχοι, ε, ακτοφυλακοί, ε, οργανισμοί δίωξης του οικονομικού εγκλήματος. Και ήθελα να χαιρετήσω σήμερα και την Ιταλική δίωξη οικονομικού εγκλήματος που σήμερα έχει την γιορτή της. Αλλά ταυτόχρονα και μη κυβερνητικέ οργανώσει υπεύθυνε για την υποδοχή, υπεύθυνε του ιατροφαρμακευτικού κλάδου, όσοι βοηθούν τα παιδιά. Ευχαριστώ λοιπόν για την φροντίδα και μέρημνα που δίνεται κάθε μέρα στους ανθρώπους αυτούς. Η συζήτηση σήμερα έχει ένα σκοπό, να κάνει να ακουστεί ε, ξεκάθαρα και δυνατά η δική σας φωνή, η δική μας φωνή, απευθυνόμενοι και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που αύριο και μεθαύριο θα συναντηθούν για να ασχοληθούν με το θέμα της μετανάστευσης. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ξεχνάμε ότι οφείλουμε να δράσουμε γοργά και με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν είναι απλή. Ωστόσο, οι πολίτες τρέφονται προς την Ευρώπη για να λύσει τα προβλήματα. Αυτό λέει το Ευρωβαρόμετρο ζητά από τα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα προβλήματα, την μετανάστευση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ανεργία των νέων, δηλαδή την κοινωνική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουν. με την κατάσταση είναι επιδεινώνεται με τον πόλεμο στη Συρία. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία. Δυσχερίες έχει και η Βόρεια Αφρική, το ίδιο και η Ποσαχάρη Αφρική. Έχουμε τη χαρά να προσκαλέσουμε και τον Πρωθυπουργό Αλ Σαράι, τον Πρωθυπουργό της Λιβύης και τον ευχαριστώ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Και θα μπορέσει να προσφέρει τη μαρτυρία του για το πόσο είναι δύσκολο να επιληθούν και τα εσωτερικά προβλήματα των διαφόρων κρατών της Αφρικής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να παύσουμε την εμπορία ανθρώπων, γυναικών και παιδιών από εγκληματικέ οργανώσεις, από εγκληματίες που κερδίζουν εκμεταλλευόμενοι την απελπισία γυναικών. Ε, αυτές που με τα παιδιά τους στα χέρια, οι μητέρες προσπαθούν να ε, ζήσουν την ελπίδα τους να ξεφύγουν από τις χώρες τους χώρες από τις οποίες φεύγουν ε, λόγω των κλιματικών αλλαγών. Η έρημος έχει καταλάβει εκτάρια επί εκταρίων ζωτικού χώρου ή λόγω του Μπόκο Χαράμ ή λόγω του λοιμού ε, και της πείνας ή λόγω των ε, φιλετικών διαφορών. Είναι άνθρωποι που θα ε, προσπαθήσουν από τον Νότο να έρθουν προς το Βορρά γιατί έχουν χάσει την ελπίδα τους. Η οργή λοιπόν και η απελπισία διωγγώνονται. Πέρα από αυτό το δράμα που ανησυχεί και τους συμπολίτε μας, η Ευρώπη δεν μπορεί να παρουσιάζεται αδύναμη ή αδιάφοροι. Εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις, οι σιρήνες του λαϊκισμού θα εκμεταλλευτούν ε, την ε, περιφρόνηση, την απόρριψη και τον φόβο και ε, δεν θέλουμε να έχουμε την αυταπάτη ότι μπορούμε να κλειστούμε πίσω από τείχη και σύνορα κλείνοντα τι πόρτε μα. Πρέπει να βοηθήσουμε του Ευρωπαίου συμπολίτε μα προσφέροντα χειροπιαστέ λύσει. Επενδύοντα και περισσότερο. Γι' αυτό είπα πολύ ξεκάθαρα ότι δεν ε, ήθελα να σταθώ σε συγκεκριμένου τομεί τη οικονομία. Όμω, ο επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασιστεί σε πολιτικέ επιλογέ. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στι επίγουσε ανάγκε του φαινομένου τη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα δημόσια τάξη και ασφάλεια. Είναι ένα πρόβλημα πολιτικό ε, ουσιώδου σημασία, κέρια σημασία που οφείλουν να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει άοκνες προσπάθειες για να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα των ε, προσφύγων. Μέρος του μεγαλύτερου ε, προβλήματος και φαινομένου της μετανάστευσης. Απειλούνται ανθρώπινες ζωές, απειλούνται οι δικές μας θεμελιώδεις αξίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δείξουμε ε, ε, την απαραίτητη πυγμή στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Όμως το τωρινό σύστημα κατανομής των προσφύγων έχει αποτύχει. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια αιτήσει ασύλου, 2,5 εκατομμύρια μόνο μεταξύ 2015 και 2016. Με τους ισχύοντες κανόνες, η Ιταλία και η Ελλάδα, οι χώρες της ε, πρώτης άφηξης, πρέπει να διαχειριστούν το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων. Είναι βαθιά ε, αδικία αυτή. Να αφήνουμε ένα τόσο μικρό αριθμό κρατών να χειριστούν αυτή την ευθύνη. Πέραν τη δέσμευση που έχουν και ε, του καθήκοντο να ελέγχουν την Μεσόγειο και να διασώζουν ανθρώπινε ζωέ στη θάλασσα. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλησαν οι ιδρυτέ τη. Η αλληλεγγύη ήταν το θεμέλιο της ε, ευρωπαϊκή συνύπαρξη. Όμως θα είτο, θα είτο ε, σφάλμα να κατηγορήσουμε για, αυτό το, ε, μεγάλο, για αυτή τη μεγάλη αδικία ε, την Ευρώπη. Αδιακρίτως το Συμβούλιο και γι' αυτό ευχαριστώ και την πρωτοβουλία του κ. Γιούνκερ πρότεινε μια μεταρρύθμιση πολύ τολμηρή η Επιτροπή για τι Ελευθερίε των Πολιτών, τη Δικαιοσύνη και τι Εσωτερικέ Υποθέσει επεξεργάζεται την πρόταση αυτή προσπαθώντα να κάνει το σύστημα του σύλλογου πιο αποτελεσματικό. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται μέχρι το τέλο του καλοκαιριού. Η μεταρρύθμιση αυτή προβλέπει ε, αυτομάτω να αναδυναμηθούν οι αιτήσει ασύλου μεταξύ των χωρών, ιδίω όταν υπάρχει πλεόνασμα σε κάποια χώρα, και να γίνουν ομογενή τα κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, προσφέρεται άσυλο. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού, εντατικότερα, για να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες. Πραγματικά εκτίμησα την ε, ξεκάθαρη επιλογή της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε μια επιπαραβάση διαδικασία εναντίον των χωρών που δεν σεβάστηκαν την συμφωνία. Ο σκοπό δεν είναι να τιμωρήσουμε κανέναν ή να επιβάλλουμε κυρώσει. Είναι απλώ να θυμίσουμε ότι τα συμφωνηθέντα, τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. Η αλληλεγγύη ε, πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και πρέπει επίσης να είναι ε, δεδομένο ότι υπάρχει δούνε και λαβίν. Θα πρέπει να ε, αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα. Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτές οι διαδικασίες επί παραβάση και ποτέ δεν ήμουν ε, θειασότη του. Όμω, όταν υπάρχουν καθήκοντα και υποχρεώσει, λογικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι θεματοφύλακα των συνθηκών, να, καλεί, να καλεί να τηρούνται οι συνθήκε και οι κανόνε. Ε, κύριε Γιούνκερ, το κείμενο ε, αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο κατά μεγάλη πλειοψηφία ε, σας στηρίζει στην προσπάθεια να κάνετε τους κανόνες σεβαστούς. Δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Υπάρχει μια σύγχυση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν κάνουν τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θέλουν να δράσουν. Τα κράτη-μέλη δεν είναι αυτά, που, είναι αυτά που δεν δρούν. Αυτά δεν σέβονται τι υποχρεώσει του. Πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα. Αυτό του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Είναι αλήθεια. Οι παραμεθόμενε χώρε υποφέρουν περισσότερο από άλλε, γιατί έχουν μεγαλύτερα βάρη και καθήκοντα σε σχέση από αυτού που δεν έχουν εξωτερικά σύνορα. Η κουβέντα αυτή μπορεί να γίνει για την Ουγγαρία, ε, αλλά σαφώς για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία. Πρέπει να προσπίζονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα, πρέπει να τα προσπιζόμαστε καλύτερα. Η ευρωπαϊκή επιλογή, όπω προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει ευρωπαϊκή ε, είναι σημαντική. Ήδη ξεκίνησε να εκδιπλώνει τη δύναμη αυτή στην ε, Ουγγαρία. Δεν μπορούμε να αφήνουμε μόνη της ε, μία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι σαφές. Και αυτή είναι μία πορεία την οποία πρέπει να την ε, συνεχίσουμε, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών. Ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος μπορούν να μας βοηθήσουν ε, σε αυτό το σκοπό. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τα εξωτερικά σύνορα, αλλά εσωτερικώς πρέπει να ενισχύσουμε και την ενιαία μας αγορά. Ε, τα ισχυρά εξωτερικά σύνορα σημαίνουν ότι τέσσερι ελευθερίε μπορούν να ασκούνται ελεύθερα. Πρέπει να, να ενισχύσουμε τα ε, εξωτερικά όμω σύνορα, όχι τα εσωτερικά, διότι αν κλείσουμε τι πόρτε μα, αυτό θα σημαίνει ότι δεν ενισχύουμε την καταπολέμηση της μετανάστευση, αλλά θα δυσκολέψουμε την εξέπρεση λύσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε αποφεύγοντας τις ουρές βεβαίως φορτηγών και ταλικών στα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να το φροντίσουμε και αυτό. Ε, φίλοι, συνάδελφοι, αγαπητέ Ζαν είναι σημαντικό να έχουμε μια πραγματική στρατηγική για την Αφρική. Η Αφρική θα πρέπει να είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα και για τα ερχόμενα χρόνια. Συμμερίζομαι πλήρω τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που προτείνει να επενδυθούν περισσότερα. Ήδη προβλέπεται ένα πακέτο επενδύσεων που υποβλήθηκε από τον αρμόδιο επίτροπο 40 δι ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διπλασιάσει τις επενδύσεις στην Λιβύη. Περάσαμε στα 400 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Πιστεύω ότι ο επόμενο ε, ευρωπαϊκός προπολογισμό και ε, με βάση την πρόταση της Επιτροπής που στηρίζεται από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να ευνοήσουμε την ανάπτυξη, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στην ίδια την Αφρική και να ε, αποφύγουμε οι νέοι, οι γενιές του μέλλοντος στην Αφρική, να χάσουν την ελπίδα, την ελπίδα ότι μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ζουν πιο ελεύθερα με αξιοπρέπεια έχοντας επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, που δίνουν μια προοπτική στους νέους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε να δούμε την Αφρική όχι με τα γυαλιά της Ευρώπης και μέσα από την δική μας οπτική γωνία, αλλά με την οπτική των Αφρικανών ε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Αφρικανική Ένωση, ο Μουσαφάκη, ε, και ο πρόεδρος της ακτής του Ελεφαντος του Αλασάνε Ουατάρα έχουν συζητήσει με το κοινοβούλιο μας. Ήδη σήμερα με την παρουσία του κυρίου Αλσαράη έχουμε πρόεδρο από το Κοινοβούλιο της Οικονομικής Κοινότητας των κρατών της ε, Δυτικής Αφρικής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την επιχειρηματική μας τεχνογνωσία, ξεκινώντας από μια ρωμαλαία διπλωματική προσπάθεια σε επίπεδο οικονομικό, πολιτιστικό και ακαδημαϊκό. Κύριε Γιούνκερ, συμφωνώ με το, για το πόσο σημαντικό ρόλο πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή διπλωματία στην προσπάθεια επίλυσης των αφρικανικών προβλημάτων. Ναι, μπορούμε να έχουμε κοινοπραξίε. Ναι, μπορούμε να στηρίξουμε τι μικρομεσαίέ επιχειρήσει. Ναι, μπορεί να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπου της Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων για τι προσπάθειε τους. Χρειάζεται μια πραγματική ε, σφαιρική στρατηγική, ολιστική στρατηγική. Είχε δίκιο ε, ο Ζαν Κλόντα όταν ανέλαβε ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι χρειάζεται πολιτική. Χρειάζεται πολιτική, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να είναι σκέτη γραφειοκρατία. Πρέπει να είναι κυρίω πολιτικού χαρακτήρα. Και η πολιτική απαιτεί και μια, τη χάραξη μια πορεία. Πιστεύω ότι η πορεία αυτή, σε ό,τι αφορά την Αφρική και την ανάπτυξη τη Αφρική, με την παρουσία όλο ένα και περισσότερο Ευρωπαίων στην Αφρική, όχι για μια νέα απεικιοκρατία στην Αφρική, όπως λένε κάποιοι, αλλά για να υπάρχει με την Ήπειρο αυτή μια σχέση ισοτήμων προς ισοτήμους. Μια αδερφική σχέση. Αδέρφια που καταλαβαίνονται καλύτερα. Άνθρωποι και λαοί που έρχονται από μακρινές Υπήρους. Εύχομαι οι προτάσεις τις οποίες τώρα συζητούμε, τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τις εγκρίνουμε με μια ευρεία συνένεση και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, Αφρικανική Ένωση, που θα γίνει στην ακτή του Ελεφαντοστού, στο Αμπιτζάν, ε, μέσα στο καλοκαίρι μάλλον στα τέλη Νοεμβρίου. Ήδη στι 25 Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, υπέγραψαν μια επίσημη δήλωση για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωση στη Ρώμη. Η βασική προτεραιότητα της Ένωσης θα ήταν ακριβώ η εξέβρεση λύσεων στο πρόβλημα της μετανάστευση Αύριο οι ίδιοι που προσυπέγραψαν αυτές τις ε, δηλώσεις θα συναντηθούν αύριο και θα πρέπει να επαναλάβουν την ανάληψη αυτής της πολιτικής ευθύνης που είναι και έκφραση πολιτικής βούλησης. Στην έναρξη λοιπόν αυτής της ε, διάσκεψης ε, στάθηκα στην σημασία ανάγκης να στηρίζεται αυτό το μήνυμα. Πρέπει να αποφασίσουμε, πρέπει να δώσουμε χειροπιαστές απαντήσεις στους ε, συμπολίτες μας. Οι πολίτες μας ζητούν μια ένωση που να είναι σε θέση να τους προστατεύσει και να ε, βεβαιώσει τις αξίες τις οποίες θεμελιώνεται. Όχι μόνο στα λόγια, στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Γι' αυτό στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι και η δική σας δράση είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ήδη είναι πολλά τα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι πρέπει να δούμε με μια προοπτική αισιόδοξη την Αφρική και να τους δώσουμε και εκείνον μια προοπτική. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι χιλιάδε πρόσφυγε που μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη, είναι τα εκατομμύρια ε, άνθρωποι που για όλου του λόγου που προανέφερα θα μπορούσαν τα ερχόμενα χρόνια να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν την Αφρική γιατί είναι απελπισμένοι και να στρέψουν το βλέμμα του προ το βορρά. Γι' αυτό πρέπει να παρέμβουμε, να δράσουμε ήδη σήμερα. Πρέπει να ε, ε, έχουμε αυτήν την ολιστική, τη σφαιρική στατικική. Είμαι πεπισμένο ότι ο Ιτζάν Κλοντ Γιούγκερ, στον οποίο θα δώσω το λόγο, μαζί μου θα φανεί ένας βασικός υπερασπιστής των πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα κοιτάζοντας με ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή την Αφρική, τη σταθεροποίηση στην Μέση Ανατολή, τη σταθεροποίηση στον χώρο της Μεσογείου και προσπαθώντας να βρούμε χειροπιαστές απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών μας, αλλά και για να αποστείλουμε ένα μήνυμα προς τους συνομιλητές μας από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Το μήνυμα αυτό να λέει ότι η Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι και θέλει να είναι φίλος ήταν, είναι, θα είναι και θέλει να είναι ένας έμπιστος πολιτικός εταίρος με τους οποίους μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον, της, ε, ε, ένα μέλλον αισιόδοξο για τα παιδιά της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Eh, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Αντώνιο, κύριε Πιτέλα, κυρία Τσίμερ. Κυρίες και κύριοι υπουργέ, ε, βουλευτές, ε, δυστυχώς δεν μπορώ να εκφραστώ στη μητρική μου γλώσσα τα λεξιμβουργιανά, γιατί μόνο λίγοι από εσάς είσαστε γνώστες της γλώσσας αυτής. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λοιπόν στις τρεις άλλες γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούμε γερμανικά. Θα ξεκινήσω με τα γερμανικά. Κυρίε και κύριοι, καταρχάς, για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε ο τίτλος ε, Ευρωπαϊκή αμα, Διαχείριση Συνόρων. Ένα πρόγραμμα σε έξι πανεπιστήμια και σε διάφορες υπηρεσίε. Ε, υπηρεσίες ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει ότι το γεγονό ότι υπάρχει πλέον αυτός ο επιστημονικός κλάδος, ότι έχουμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το κοινό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε με τη Frontex καταδεικνύει ότι είναι κοινό μα καθήκον εκείνη η διαχείριση και προστασία των συνόρων μας. Μαζί με πολλούς από εσά. σε λιγότερο από ένα έτος, καταφέραμε να πετύχουμε κάτι το οποίο πριν από 20 χρόνια δεν θα ήταν δυνατόν. Να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή συνοριαφυλακή και ακτοφυλακή. Και αυτό για την ασφάλεια και την ε, φύλαξη των πιο επικίνδυνων κομματιών, ε, των πιο ευάλωτων κομματιών των ευρωπαϊκών μας ε, συνόρων στην Ελλάδα, 403 στην ε, Ιταλία, στην Ισπανία, στην ε, Βουλγαρία και επίσης έχουμε 50.000 άτομα τα οποία είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για την συλλογία φυλακή. Αυτό καταδεικνύει ότι κάνουμε ήδη ό,τι πιο σοβαρά μπορούμε για την προστασία των σύνορων μας. Στην μεταναστευτική μας πολιτική έχουμε δύο βασικές αρχές, η ευθύνη και η ελληνική. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με άλλους κατά τη διάφορα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ε, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν ε, χωρίς βοήθεια όταν βρίσκεται σε ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν να κρίνει μόνο η γεωγραφική θέση του καθενός, ε, την ευθύνη που έχει. Και θα ήθελα να επενέσω τις εξαιρετικές ε, προσπάθειες της Ιταλίας και της, Ιταλί και της Ελλάδας. Η Ιταλία δίνει ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και η Ελλάδα πράττει το ίδιο. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνοι του μόνη τη στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η Κομισιόν λοιπόν βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει τα κρατημέλη αυτά. Στην Ελλάδα και στην Ιταλία έχουμε δημιουργήσει κεντρικά κέντρα απορρόφησης τα οποία δουλεύουν ε, Ευρωπαίοι υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες από τα κρατημέλη, αποσπασμένοι. Και επίσης ε, φροντίσαμε οι ετούντες άσυλο στην ε, ε, Ελλάδα να μπορούν να διεκπαιρεθούν πιο γρήγορα αυτές οι αιτήσει 8% το 2015, ένα χρόνο αργότερα ήταν 100% η απορρόφηση αυτή. Δημιουργήσαν λοιπόν δομές, αυτές τις δομές που χρειαζόμασταν και να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει μια τακτική αντιεκπαιρέωση των αιτήσεων. Επίσης, φροντίσαμε και για τους πρόσφυγες που έρχονται μέσω επικίνδυνων οδών στην Ευρώπη. Μιλάμε για 50.000 και πλέον άτομα. Και για τον σκοπό λοιπόν αυτό υπάρχει και συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί ο αριθμός των ε, μεταναστών και των προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά. Κυρίε και κύριοι, όλα αυτά αποτελούν μια υπενθύμηση για το τι έχουμε πετύχει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο χρόνο και μόνο πάνω από 6.000 ε, άτομα έχουν έχουν ε, ε, λάβει ασφαλή τρόπο για να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν φτάνουν αυτά τα στοιχεία αλλά πρόκειται για μια ιστορική α, πρώτη φορά και έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 θα έχουμε πετύχει πολλά παραπάνω. Η ελληνική όμως δεν αποτελεί μόνο μονόδρομο. Κάθε χώρα θα πρέπει λοιπόν να κάνει αυτό που της αναλογεί ό,τι αφορά την ευθύνη της. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να έλθει στο ύψος των περιστάσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, με, τη διαδικασία, με τις διαδικασίες παραβάση τις οποίες ξεκινήσαμε καταδείξαμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τις ευθύνε μας. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι κάτι που με ικανοποιεί να ξεκινούμε διαδικασίες επί παραβάση. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορώ να πείσω. Διότι η αλληλεγγύη πρώτα έρχεται από την καρδιά. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να πάρουμε μέτρα για να γίνουν σεβαστές δεσμευτικές αποφάσεις. Και πρέπει βεβαίως το σύστημα για το μέλλον ε, να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Οι διαδικασίες είναι περίπλοκες, είναι μακροσκελής και οι αιτούντες άσυλο δεν είχαν τις ίδιες μεταχείρισης σε όλες τις χώρες. Κάποια συστήματα ασύλου είναι πιο γενναιόδωρα από άλλα. Και αυτό βεβαίως ενθαρρύνει την επιλογή τόπου ασύλου. Και βεβαίως το παρόν σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει υποπίεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ισχυρό σύστημα που θα βοηθάει τα κράτη-μέλη που πλήττονται περισσότερο γεωγραφικά και θα προστατεύει όσους δεν έχουν που αλλού να πάνε. Αυτή ήταν η βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του, συστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Οι προτάσεις μας εγγράφονται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και προσπαθούμε αυτό να το σε όλες τις πτυχές, από τις συνθήκες ε, υποδοχής, ε, την επεξεργασία των μετήσεων ασύλου, την κατανομή ευθυνών, Θέλουμε να εναρμονίσουμε τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μην έχουμε δευτερογενεί μετακινήσει και, και επιλογή τόπου ασύλου. Και βεβαίω ταυτόχρονα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι καταχρήσει και τι τρευλώσει. Πιέζει ο χρόνο και πρέπει να προχωρήσουμε. Χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωράει σταθερά προ την κατεύθυνση αυτή. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Μαλτέζικη Προεδρία, αλλά και τη μελλοντική, την Εσθονική και την προηγούμενη τη Σλοβάκικη για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το διέξοδο. Πρέπει ήρθε η ώρα να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό ισορροπημένο έτσι ώστε το σύστημα ασύλου να μπορεί να εξυπηρετήσει το σκοπό του. Κυρίε και κύριοι, όταν μιλάμε για μετανάστευση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία, πίσω από του αριθμού, υπάρχουν γυναίκε, άντρε, παιδιά που θα προτιμούσαν να είχαν μείνει στο σπίτι τους αντί να πάρουν τους δρόμους για να αποφύγουν τον πόλεμο, τη βία και τη φτώχεια. Είναι δική, δική μας ευθύνη, δική μας των Ευρωπαίων, οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον στις δικές τους χώρες, αντί να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους στη Μεσόγειο και να πλουτίζουν οι διακινητές. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία μας με τις χώρες προέλευσης και τράνζιτ όπως ε, πολύ σωστά υπογράμμισε και ο Πρόεδρος με τους Αφρικανούς ξαδέρφους μας. Πέρυσι ξεκίνησε ε, ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με την ε, Αφρική. Ενισχύθηκε η καταπολέμηση των διακινητών με την ενίσχυση των, της ακτοφυλακής της Europol και με την αποστολή Σοφία στη Μεσόγειο όλοι όσοι συμμετέχουν σε όλο, όλα αυτά τα όργανα ε, πραγματικά αξίζουν συγχαρητηρίων και όσοι συμμετέχουν στην Αποστολή Σοφία καθώς και όσοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Ακτοφυλακής ε, και Συνοριοφυλακής ε, έχουν κάνουν μια δουλειά αξιοσημείωτη χωρίς αυτούς θα ήμασταν χαμένοι και θα χανόντουσαν και πολλοί ακόμα δύστοιχοι άνθρωποι έχουν παρθεί μέτρα για να διευκολύνουμε την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στη χώρα προέλευσής τους. Τα προγράμματα ενίσχυσης, ε, τα οποία ξεκίνησαν από την ε, Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης με την υποστήριξη την οικονομική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη επέτρεψε σε πάνω από 4.000 μετανάστες που ήταν μπλοκαρισμένοι στη Λιβύη να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους και οι συμφωνίες επανεισδοχής βρίσκονται διαπραγμάτευση με το Μαρόκο, την Τινησία, την Ιγυρία και την Ιορδανία. 200 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν ε, το 2017 για δράσεις ε, που αφορούν τη μετανάστευση στη Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, αλλά και στην Αίγυπτο και την Τινησία. Επίσης, το επίγον ταμείο για την Αφρική έχει κινητοποιήσει 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν εγκριθεί πάρα πολλά project με, την, με τον Ήγυρα, τη Σενεγάλη, αλλά και το Νότιο Σουδάν. Επίσης υπάρχει και ένα πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων για την Αφρική και τις γειτονικέ χώρες. Και ελπίζω οι συνομοθέτες να κινηθούν γρήγορα, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να μπορέσει να είναι επιχειρησιακό σύντομα. Έχουμε γράψει πολλά ποίηματα, έχουμε πει πολλά για τη συνεργασία με την Αφρική. Πρέπει όμως τώρα να επενδύσουμε εκεί, επιτόπου στην Αφρική, για να μπορέσει και η Αφρική να είναι παρούσα ε, όταν προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της και τις φιλοδοξίες της. Ε, έχουμε κάνει πολλά για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα μεταναστευτικά ζητήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι όμως ε, η ώρα για να συγχαίρουμε τον εαυτό μας και να επαναπαυόμαστε. Πρέπει να συμπληρώσουμε, πρέπει να ενισχύσουμε τα, τη βάση την οποία έχουμε δημιουργήσει. Είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχουν γίνει. Έως τώρα, ναι και όχι. Μένουν πολλά να γίνουν και θα τα κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητέ Ζαν Κλόντ, για την ομιλία σου και για την υποστήριξή σου ε, γενικότερα του όλου εγχειρήματο. Ιδιαίτερα γιατί έχεις δεσμευτεί σε αυτόν τον τομέα και μπορείς να βασιστείς στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη, και καταρχήν θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την εργασία της τόσο στην Αφρική όσο και αλλού για να δοθούν και να βρεθούν λύσεις. Να βοηθήσουμε εκείνους που φεύγουν από τα σπίτια τους στην υποσαχάρια περιοχή. Και για εκείνους που φεύγουν από τη χώρα τους λόγω της τρομοκρατίας, ε, του λοιμού και της απερίμωσης. Γι' αυτό έχουν δεσμευτεί όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ Αντώνιο, θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου, θα μιλήσω Ιταλικά τη στιγμή που υπάρχει ε, διερμηνία και, εν πάση τα Ιταλικά ε, ομιλούνται λίγο περισσότερο από τα Λουξεμβουργιανά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνιο για τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης σήμερα με τη συμμετοχή τόσων εταίρων που συνεργάζονται μαζί μας για την διαχείριση ενός δύσκολου φαινομένου. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση κατεπήγοντος μόνο, θα πρέπει να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα ε, δύσβατο ζήτημα. Γι' αυτό χαίρομαι για το γεγονός ότι παρευρίσκονται εδώ και πολλοί διεθνείς εταίροι. Γιατί τα τελευταία δυόμιση χρόνια, αν καταφέραμε κάτι, το καταφέραμε και με την συνδρομή των διεθνών εταίρων μας. την ημέρα πριν από την ακρόαση που είχε διοργανωθεί τις 3 Οκτωβρίου το 2014 ήμουν στη Λαμπεντούζα και είχα υπενθυμίσει ποια ήταν τα θύματα αυτής ε, της μεγάλης τους πορείας προς την απώλεια. Και βεβαίως αυτό το είχαμε τονίσει και με τον Ζαν Κλοντ. Μιλήσαμε για την τροπή που αισθανόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κλείσαμε τα μάτια μας προς τις χιλιάδες νεκρών που έρχονται στη δική μας θάλασσα και αυτούς που κινούνται από την υποσαχάρια περιοχή, από το Σαχέλ και έρχονται προς τη Μεσόγειο. Εγώ είχα εκφράσει την ντροπή μου για τους νεκρούς που τόσα χρόνια κάναμε ότι δεν βλέπαμε. Και χαίρομαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση που σώζει ζωές στη θάλασσα και νομίζω ότι κάθε ζωή που δεν διασώζεται αποτελεί ήττα για μας. Τα τελευταία δυόμιση ε, χρόνια είχαμε μεγάλες απώλειες, όπως είπε και ο Ζαν Κλοντ και ο Αντώνιο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τη μεταναστευτική πολιτική είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αρχικά ήταν θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών. Νομίζω ότι καταφέραμε μαζί να το επιτύχουμε αυτό. Δηλαδή, όποιος έρχεται στην Ευρώπη, έρχεται στην Ευρώπη και όχι σε μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη από τα θεσμικά όργανα, τα κράτη και τους πολίτες στο σύνολό τους. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο, ιδιαίτερα ως προς την εσωτερική αλληλεγγύη, όπως τόνισαν και ο Αντώνιο και ο, Ζαν Κλοντ. Και είναι και θέμα εξωτερικής ευθύνης που έχουμε αναλάβει. Όταν συνειδητοποίησα ότι το θέμα αυτό δεν ε, βρίσκεται στην ατζέντα των ε, Υπουργών Εξωτερικών, κατάλαβα ότι το θέμα είχε προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται μία συντονισμένη δράση εξωτερικής πολιτικής με βάση την Ένωση αλλά και τη διαφορετικότητά μας. Έχουμε προβάλει πέντε δράσεις τα τελευταία δυόμιση χρόνια μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Με μία ένωση, ενότητα ως προς την αντιμετώπιση, ως προς τα εξωτερικά σύνορα, γιατί ως προς την εσωτερική δράση έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο. Καταρχήν μας ενδιαφέρει να σώσουμε ζωές στη θάλασσα αλλά και στην ε, έρημο γιατί βλέπουμε τη θάλασσα, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς είχαν τη ζωή τους στην έρημο της Αφρικής την προηγούμενη εβδομάδα. Με τις αρχές του Νίγηρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη σώσαμε 100 ζωές, γυναίκες και παιδιά που είχαν εγκαταλειφθεί στην έρημο χωρίς νερό και χωρίς φαγητό. Και με βάση την ε, συνδρομή του Νίγηρα σώσαμε ζωές και προβάλαμε και μία εναλλακτική για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Μόνο η ακτοφυλακή της Λιβύης έσωσε 23.000 ανθρώπους μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης Σοφία. Έτσι ώστε οι Λίβοι να μπορέσουν να ασκήσουν έλεγχο στα χωρικά τους ύδατα, δηλαδή να σώσουν ζωές, αλλά να μπορούν να έχουν και ελεύθερη δράση και οι αλλοί της περιοχής. και είναι δεκάδες, χιλιάδες οι ζωές που ε, σώσαμε. Όποιος από εσάς μίλησε με μία γυναίκα η οποία επιβιβάστηκε σε ένα φουσκωτό με τα παιδιά της έγκυος και ήθελε να διασχίσει τη Μεσόγειο, ήξερε τι διακινδυνεύει και αν το διακινδυνεύει σημαίνει ότι αυτή η όθηση δικαιολογείται. Θα πρέπει να διασώσουμε ζωές και έχουμε διασώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Και όχι μόνο να διασώσουμε αλλά και να προστατεύσουμε. Είμαι υπερήφανη γιατί μαζί με την Διεθνή Οργάνωση μετανάστευσης και με τους φίλους από τη Λιβύη καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα κράτησης στη Λιβύη όπου οι καταστάσεις διαβίωσης είναι δραματικές και μόνο οι διεθνείς οργανώσεις μετανάστευσης μπορούν να εγγυηθούν καλύτερη διαβίωση και αυτό αφορά και την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί όταν συνεργαζόμαστε, τότε δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και μπορούμε να οδηγηθούμε και σε επιστροφές. Γιατί πάνω από 400 πάνω από 450.000 επιστροφές ε, διασφαλίστηκαν. Και αυτό με βάση τη συνδρομή και της Λιβύης. Και με βάση αυτή την εταιρική σχέση προσπαθούμε να προωθήσουμε τις επιστροφές στον Ήγηρα το ίδιο. 2.600 άνθρωποι τους τελευταίους μήνες επανήλθαν στη χώρα προέλευσης με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Μας ενδιαφέρει επίσης η διάσωση των ανθρώπων και η καταπολέμηση των διακινητών. Μέσα στα πλαίσια και τις επιχείρησης Σοφία καταφέραμε να συλλάβουμε πολλούς διακινητές, 500 σκάφη τα εξουδετερώσαμε, αλλά και στις χερσαίες επιχειρήσεις στην Αφρική, δύο εβδομάδες πριν, καταφέραμε μεταξύ των πρώτων εταίρων να δώσουμε 50 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή του Σαχέλ έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να ελέγχουν τον τόπο τους κατά των διακινητών και των λαθρεμπόρων. Αυτό προωθούμε εταιρική σχέση, ενίσχυση των εταίρων μας και καταπολέμηση της τρομοκρατίας επιτοπίως. Τέταρτον, θα πρέπει να άρουμε τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτή τη φύγη. Ο Αντώνιο έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να γίνει να γίνουν μαζικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της Αφρικής ε, από οικονομικής, κοινωνικής ε, πλευράς, καταπολέμησης της τρομοκρατίας, κλιματικών αλλαγών και ούτω καθεξής. Είναι όλοι παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να συνδράμουμε. Γιατί εμείς είμαστε η γειτονική Ήπειρος. Κανένας δεν είναι πιο κοντά στην Αφρική. Μιλάμε για βόρεια και νότια όχθη της Μεσογείου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις γεωγραφικές μας παραμέτρους. Όταν μιλάμε ας πούμε για την Μάλτα και ξέρουμε πόσο κοντά είναι στην Τινησία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα προωθήσουμε. Εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και όχι ένα σχέδιο Marshall. Ιδιωτικές επενδύσεις μαζί με εξωτερικές επενδύσεις, μια συνέργεια με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα βοηθήσουν τις ευάλωτες αφρικανικές χώρες με τις αντιπροσωπείες μας επιτοπίως και βεβαίως και κοινωνική ανάπτυξη, δημοκρατική ανάπτυξη περιβαλλοντική ανάπτυξη αλλά και ψηφιακή στην Αφρική. Είναι κοινή μας ευθύνη. Και αυτό είναι και το τελικό σημείο. Έχουμε προωθήσει εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες προέλευσης των μεταναστευτικών ορών. Μιλάμε για σύμφωνα, για compact. Ήταν ευρωπαϊκή η ιδέα και ήταν πολύ καλή και τα Ηνωμένα Έθνη συνδράμουν. Είναι η λογική της εταιρικότητας. Δεν υπάρχει βοράς κατά του νότου ή τούμπαλιν, αλλά ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε με την εσωτερική μας αλληλεγγύη, στη Μεσόγειο επίσης με τη συνεργασία με τις γείτονες χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου, με την Αφρική που είναι η πιο γειτονική μας Ήπειρος, αδελφή Ήπειρος και με τα Ηνωμένα Έθνη, με τη σύνδρομή τους. Έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις πολύ σχέσεις. Δεν μιλάμε μόνο για έλεγχο των συνόρων, μιλάμε για ανάπτυξη, για βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο Αγκαντές βορείως του Νίγηρα η πύλη, από την πύλη εισόδου προς τη Λιβύη είχαμε 70.000 διελεύσεις. Φέτος είναι 5.000 οι διελεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο σοβαρής εργασίας καταφέραμε να μειώσουμε άρδιν τους αριθμούς. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά βρισκόμαστε στη σωστή οδό και νομίζω ότι με τη συνδρομή όλων των θεσμικών οργάνων θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φεντερίκα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Πρωθυπουργό της ε, Λιβύης, τον Αν Σαράι. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για αιτήματα, ανάγκες και προβλήματα μίας από τις βασικότερες χώρες που θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Μία χώρα που υποφέρει, που καταβάλει προσπάθειες και που είναι πρωταγωνιστής για να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός Αλσαράζ. فخامة السيد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو Ταϊάνι. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Αντώνιο Ταγιάννη, κυρίες και κύριοι εξοχότητές σας. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Αντώνιο Ταγιάννη, για το γεγονό ότι μα κάλεσε σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερω για το θετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ε, κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης προκειμένου επιτέλους να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη στην αγαπημένη μου χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προσπάθειες που καταβάλει για να συνεργαστεί με τη χώρα μου σε όλους τους τομείς και όλους ιδιαιτέρως ε, ευχαριστώ την Ιταλική κυβέρνηση η οποία τον τελευταίο καιρό μας παρέχει άμεση βοήθεια και υποστηρίζει διάφορα προγράμματα για την καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης ε, και πέραν τούτου μας υποστηρίζει σε πάρα πολλά ε, τμήματα των εργασιών μας στη Λιβύη. Κυρίες και κύριοι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μου στην παρούσα φάση, καταβάλουμε προσπάθειες να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και τις συνέπειε. Υπάρχει η ανθρωπιστική διάσταση, η διάσταση τη ασφάλεια, αλλά και η οικονομική διάσταση. Οι πρόσφυγε λοιπόν θα πρέπει να τη χάνουν ανθρώπινη ανθρώπινης θα πρέπει να, έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρέπεια, δεδομένη και τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξασφαλίσουμε και επίσης το πρόβλημα των προσφύγων και της μετανάστευσης δεν μπορούμε να το επιλύσουμε μόνο με θέματα ασφάλειας. Οι χώρε από τι οποίε προέρχονται οι μετανάστες είναι χώρε τι οποίε πρέπει να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση αλλά και η όροι διαβίωση των πολιτών στι χώρε αυτέ, καθώ και να υπάρξουν ευκαιρίε για απασχόληση των νέων. Και κυρίω λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιταλία και την Γερμανία γιατί δημιούργησαν α, προγράμματα υποστήριξης και ανάπτυξης της χώρες ε, από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες κυρίως στη χώρα μου και αυτό είναι κυρίως ε, στα νότια σύνορα. Εκεί λοιπόν πλέον μπορούμε να επιβάλλουμε να, πιο πολλά μέτρα ασφάλειας. Ε, κυρίες και κύριοι, η Λιβύη είναι χώρα από την οποία περνάνε πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες και μας αυτό το πρόβλημα εξίσου όπως και την Ευρώπη. Ξέρουμε πόσο αρνητικές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις για όλους τους τομείς της ε, ζωής. Δημιουργεί επιβάρυνση την οποία η Λιβύη δεν μπορεί να σηκώσει μόνη τη και δεδομένου του προορισμένου προϋπολογισμού που έχουμε για την ανάπτυξη, για την καταπολέμηση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ήταν πολύ αρνητικέ οι συνέπειε. Υπήρξαν ξέσπασμα ασθενειών, εγκληματικών δραστηριοτήτων, τρομοκρατικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι μέσω των μεταναστευτικών αυτών κυμάτων κατέφτασαν στη χώρα μας. Και επίσης ήταν πάρα πολλές οι ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάθηκαν στη χώρα τον τελευταίο καιρό λόγω των προβληματικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Παρά τι αρνητικέ συνέπειε των μεταναστών για τη ζωή στη χώρα μου και για το νότιο τμήμα της χώρας μου, κυρίες και κύριοι. 4.000 χιλιόμετρα είναι τα χερσαία σύνορα μας και 2.000 τα θαλάσσια σύνορα της Λιβύης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να φυλαχτούν αυτά τα σύνορα και προς την κατεύθυνση αυτή χρειαζόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα μέσα αλλά και ιδιαίτερε προσπάθειε. Αυτά τα μέσα λοιπόν δεν τα έχουμε στην παρούσα φάση στη διάθεσή μα. και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υποδείξω ένα πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23, 23 ε, Ιου, Ιουλίου του 2016. Με τα ευρωπαϊκά λοιπόν αυτά μέσα, στο νότιο τμήμα της χώρας μας, ε, θέλαμε να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, γιατί στο νότιο τμήμα ξεκινάνε τα ζητήματα και εκεί φυσικά είναι και το θέμα της συνεργασίας με τα κοινά σύνορα, με τις ε, γειτονικέ μας χώρες. Αυτά τα κοινά σύνορα λοιπόν σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Πριν από δύο εβδομάδες και επισήμω καταθέσαμε έτοιμα στον ΟΗΕ για την άρση του εμπάρκου στη Λευκή Ακτή προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Και προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Εθνική Κυβέρνηση Συμφιλίωσης ασφαλώς προσπαθεί να δώσει τα απαραίτητα σε αυτούς που βρίσκονται στην ε, επικρατειά μας μέχρι ότου επιστρέψουν στη χώρα τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν κορυφαία προτεραιότητά μας και γι' αυτό είναι λοιπόν τόσο σημαντικό να κλείνουμε συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης προκειμένου να μην βρισκόμαστε στην κατάσταση όπου πρέπει να υποδεχόμαστε τόσους πολλούς πρόσφυγες, να χρειάζονται καταβλισμοί. Γιατί σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Θέλουμε τα εφιστάμενα κέντρα τα οποία υπάρχουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν ε, αρμόδιο είναι το Υπουργό Ιστορικών. Η συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών λοιπόν είναι κάτι το εντελώς ουσιώδες και γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε μια διεθνή συνεδρίαση υπό αιγίδα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου σε διεθνές επίπεδο να εξετάσουμε το θέμα αυτό και τις αρνητικές συνέπειες ε, του προβλήματος, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ε, μέσω της χώρας μου, με ό,τι συνέπειες συνεπάγεται ε, οργανωμένο έγκλημα διακίνηση ανθρώπων. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Λιβύη να το επεξέλθει στα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν οι έμποροι οι οποίοι εμπορεύονται ανθρώπινες ζωές να τερματιστεί η δραστηριότητά τους. Θα πρέπει να σταματήσει και η οικονομική τροφοδότηση των κυκλωμάτων αυτών. Και έτσι μόνο μπορούν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις μας, να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης. Έχετε δει τι υπομονή έχει επιδείξει η κυβέρνησή μας και τι θυσίες έχει κάνει η κοινωνία μας για να υπάρξει επιτέλου ε, σταθερότητα και ασφάλεια στην Τρίπολη. Η συμφιλίωση μεταξύ των διάφορων ε, περιφερειών και δήμων ε, προχωράει και έτσι ο κόσμος ξαναπηγαίνει στα σπίτια του, επιστρέφει στα σπίτια του. Και έχουμε πλέον προλιάνει το έδαφος για να σημειώσουμε τέτοιο πρόοδο. Αλλά κυρίε και κύριοι δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία Χρειαζόμαστε σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ για τη μαρτυρία σας και για την αναγνώριση που εκφράσατε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο. Να γνωρίζετε ότι η Λιβύη μπορεί πάντοτε να υπολογίζει στη στήριξη της Ευρώπης προσπαθήσουμε από κοινού να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Πριν περάσουμε στις δύο των τρογγυλής τραπέζη να δώσω το λόγο σε ορισμένους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, τους οποίους θα παρακαλέσω να τηρήσουν το χρόνο ομιλία που προβλέπεται από το Κοινοβούλιο. Είναι σύντομο ο χρόνο, αλλά έχουμε πολλούς προτεκτημένου σήμερα. Οπότε μπορούμε να δείξουμε περιορισμένη ευελιξία στο χρόνο αγόρευσης. Πρώτα απ' όλα, ο ειδικό εκπρόσωπο των ΗΕ για τη διεθνή μετανάστευση, η Λουίζα Άρμπουρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εξοχότητες, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Έχω να επενέσω το Κοινοβούλιο που ε, οργάνωσε αυτή τη διάσκεψη σε μια δύσκολη στιγμή για τη διεθνή κοινότητα, καθώς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να δημιουργήσουμε δρόμους για έφτακτη, νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με αυτό το διπλό σύμφωνο που συζητήθηκε στον ΟΗΕ. Στα πλαίσια τώρα αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να πάρω λίγα λεπτά από το χρόνο σα για να θίξω μερικά τα κρίσιμα ζητήματα που και εσεί θα συζητήσετε κατά τη διάρκεια αυτή τη διάσκεψη και που χρειάζεται να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, να δούμε τα γενεσιουργά αίτια, την αντιμετώπιση τη ε, παράνομη μετανάστευση, το πώ θα ευνοήσουμε τι επιστροφέ και θα επιτρέψουμε την ένταξη κρίση της μετανάστευσης σε διεθνές, τοπικό και εθνικό επίπεδο συνεχίζει να εκδηλήσεται, καθώς το 2017 όπως τα γνωρίζετε 2.400 γυναίκες, άντρες και παιδιά έχασαν τις ζωές τους σε μεταναστευτικές οδούς παγκοσμίως, 70% στη Μεσόγειο. Εν τω μεταξύ, καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνται ασφαλώς και νομίμως προς άλλες χώρες, ε, ταξιδεύοντας, πληρώνοντας φόρους, δουλεύοντας και κάποιες φορές επιστρέφουν και θελός στις χώρες τους. Απέναντίας κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν ε, επιλογές βασισμένες στην απελπισία, στην ε, αναζήτηση της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας σε κάποια άλλη χώρα τα κίνητρά του ε, και οι πιέσει που δέχονται στην άσκηση τη ελεύθερη επιλογή του έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα τη του. του. Ε, Κάποιε φορέ εξαναγκάζονται να προχωρήσουν, να φύγουν αλλού. Και τα αίτια είναι πολλέ φορέ ε, περίπλοκα και οφείλονται σε διαφορετικές κατηγορίες καταστάσεων. Κάποιοι είναι θύματα διώξεων, κάποιοι είναι θύματα φτώχεια, γνωρίζουν τι αντίξωε συνέπειε των κλιματικών αλλαγών ή ένα συνδυασμό των άνωθη. Γι' αυτό Μην ξεχνάμε το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι όλα τα άτομα γεννούνται ελεύθερα και ίσα ως προς τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει αυτό να το δούμε και κυριολεκτικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ε, όσο κινούνται οι άνθρωποι, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν κινούνται όλοι και θελό, αλλά μπορεί να μετακινούνται για λόγους διαφορετικούς από τα οικονομικά συμφέροντα ή λόγους. Υπάρχουν λόγοι που τους υποχρεώνουν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να σκεφτούμε τη θέσπιση κάποιων μέτρων για να διαχειριστούμε καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές και όπου χρειάζεται να προσπαθήσουμε να τις αναχαιτήσουμε, να τις συγκρατήσουμε. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον η στρατηγική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες όπως εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ε, δείχνει ότι η μετανάστευση θα πρέπει να βασίζεται στην επιλογή και όχι στην υποχρέωση. Υπάρχουν πολλά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια τα γενεσουργά αιτία τη μετανάστευση. Λόγω χάρη την ε, ε, υλοποίηση τη ατζέντα για το 2030 και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πλήρη υλοποίηση του πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά θα απαιτήσουν πολύ χρόνο, αλλά μπορεί να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την πίεση που υποχρεώνει πολλού ανθρώπου να εγκαταλείπουν τι χώρε του. Όμως η ανάπτυξη από μόνη της δεν θα ε, εξαλείψει τη μετανάστευση, ούτε θα πρέπει να είναι αυτός ο στόχος μας. Να είμαστε ξεκάθαροι ότι το Διεθνές Σύμφωνο και ο στόχος του είναι να διευκολύνει την ασφαλή, εφτακτή και νόμιμη μετανάστευση. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ε, ανάκοψη της πορείας, ούτε με την πάυση της μετανάστευσης. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ως προς τη μετανάστευση ότι υπάρχουν παράγοντες που κάποιες φορές επηρεάζουν την επιλογή του προορισμού των μεταναστών. Πολλές φορές η παραοικονομία που για πολλούς ε, μελλοντικού ε, μετανάστες ε, είναι ένας πόλος έλξης. Τώρα, η μετανάστευση, ο κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι να αυξήσουμε τους νόμιμους δρόμους για την νόμιμη μετανάστευση ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού και την ε, δυνατότητα των κρατών να ενισχύσουν τις τοπικές αγορές εργασίας και μέσω της έλευσης μεταναστών πολλές φορές. Ως το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει έλλειψη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εργαζομένων, ενώ θα υπάρχουν πολλές καινές θέσεις στον τομέα της πληροφορίας και των τεχνολογιών. Αναγνωρίζω την δυνατότητα να υπάρξει πρόσβαση σε ευέλικτες αγορές εργασίας για μετανάστες υψηλών δεξιοτήτων με το σύστημα που τώρα υπάρχει. Όμως οι ανάγκες αυτές δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στους μετανάστες υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση για την νόμιμη μετανάστευση, μετανάστευση ε, αλλάζοντας τους κανόνες για την ε, μετακίνηση και την κυκλοφορία των εργαζομένων, καθώς και για εκπαιδευτικούς ή ε, μορφωτικούς λόγους. Θα πρέπει πολλοί να πάψουν να αναγκάζονται σε παράνομους δρόμους μετανάστευσης. Υπάρχουν σαφείς ανάγκες εργατικού δυναμικού σε πολλές κοινωνίες και αυτή δεν θα πρέπει να αφήνεται στα χέρια της παρενοικονομίας. Εξοχότητες, οι επιστροφές και οι επανεισδοχές είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των συνόρων. Εκεί απαιτείται ενισχυμένη διεθνή συνεργασία. Πρέπει όμως όλα αυτά να γίνονται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια καθώς και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε μπορεί να ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε αυτή την ευθύνη. Πρέπει να γίνονται όλα αυτά με τρόπο υπεύθυνο και με νόμιμες και σωστές διαδικασίες. Οι δίκαιοι νόμοι που θα εφαρμόζονται με τρόπο δίκαιο ήταν και είναι καθοριστική σημασίας για τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και θα κρίνουν και την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Πράγματι, είναι ηρωνία ότι ε, έχει γίνει ένας τέτοιος πόλος έλξης ε, αυτό το, αυτή η Ήπειρος. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να ε, ξεχάσουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε έξω από την Ευρώπη τους μετανάστες, διότι τότε το τίμημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα είναι πολύ υψηλό, υπερβολικά υψηλό πιστεύω. Τέλος, η ένταξη και το αντιμεταναστευτικό αίσθημα στην Ευρώπη. Σημερίζομαι τις ανησυχίες ότι έχουν ε, γίνει αντιληπτοί ως ε, βάρος ή απειλή οι μετανάστες πολλές φορές και ότι κάποιοι χρειάζονται, αισθάνονται ότι χρειάζονται προστασία από αυτούς. Όμως, Τέσσερι οι προκαταλήψεις ουσιαστικά μαυρώνουν την θετική πραγματικότητα τη μετανάστευση, τη χώρε προέλευση και δυσκολεύουν τα πράγματα για τι χώρε προορισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τι προσπάθειε για την καταπολέμηση τη ξενοφοβία και να επιτρέψει την επιτυχή ένταξη των μεταναστών επιτρέποντα του να κερδίσουν τη ζωή του, αλλά και να καλύψουν ανάγκες των κοινοτήτων ε, στι οποίε βρίσκονται κοντά και εντάσσονται. Μερικές από τις πιο ευημερούσες χώρες ε, στον κόσμο έχουν βασιστεί τον εργατικό μόχθο αλλοδαπών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό να πάψει να ισχύσει σήμερα και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός αυτό και την ανάγκη αυτή. Ε, πρέπει να τηρήσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις και τις πολιτικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως απαιτεί, καθώς απαιτούνται μια προσέγγιση με συλλογικές προσπάθειες και αλληλεγγύη για την διαχείριση της μετανάστευσης εντός ε, όλων των χωρών και σε συνδυασμό μεταξύ τους και με συνεργασία με τις χώρες προέλευσης ε, από τις χώρες προορισμού. Όλα αυτά για να προωθήσουμε την κινητικότητα, την κινητικότητα των ανθρώπων με έναν τρόπο ασφαλή, έφτακτο και νόμιμο. Αν υπομονώ να συνεργαστώ με όλες και όλους σας προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άρμπουρ, για την ομιλία σας. Πρέπει απλώς να σεβόμαστε το χρόνο ομιλίας. Διότι στις 4 ο πρόεδρος Γιούνκερ θα αποχωρήσει. Και χρειάζονται και 10 λεπτά για συνέντευξη τύπου. Πολύ σύντομα λοιπόν όλοι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ο κ. Μάρκουλα. Ε, Κύριε Πρόεδρε, είπα, κυρία, είπατε εκπρόσωπε, αξιότιμη προσκεκλημένη, έχουμε την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας που μας υποχρεώνουν εδώ πρώτης ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώσουμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος της ε, διαχείρισης των μεταστικών ροών στις περιφέρειες, στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Έχουν προσκληθεί εδώ πολλοί δήμαρχοι, και μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών έτσι ώστε να μας πούν άμεσα να αναφέρουν τι συμβαίνει στις περιοχές τους. Η προσπάθεια υποδοχής, ένταξης, η καταπολέμηση του κινδύνου της ριζοσπαστικοποίησης ε, και στις ίδιες τις δικές μας κοινότητες. Μόλις επέστρεψα από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα όπου συνάντησα πολίτες αλλά και τις τοπικές κυβερνήσεις που ε, εργάζονται στα ανατολικά σύνορα πολύ εκτίθενται άμεσα από τον Δήμαρχο της Κατάνια έως τον Περιφερειάρχη της Σαλονίκης. Πρέπει να γνωρίσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Περίπου 90% αυτών των μεταναστών περνούν από τη Λιβύη και εκτίθενται στους διακινητές της εγκληματικές δραστηριότητε. Από την άλλη Υπάρχουν εξαιρετικέ περιπτώσει ό,τι φορά την Ανατολική Μεσόγειο, ε, την Τουρκία, το Λίβανο, που χρήζουν οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των κανόνων του Δουβλίνου είναι απαραίτητη. Οι πολίτε θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να προστατεύει, θέλουν ένα πιο σταθερό, πιο ολοκληρωμένο σύστημα ασύλου που θα βασίζεται στην αρχή τη αλληλεγγύη. Πολλέ πόλει και περιφέρειες επηρεάζονται άμεσα από τις μεταναστευτικές ροές. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούνται και ευκαιρίες επιτυχίας. Γι' αυτό χρειάζεται αλληλεγγύη, γι' αυτό χρειάζεται πιο έντονη διαθεσμική συνεργασία όπως προτείνει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά μένουν να γίνουν, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα των εργασιών μας στην περίπτωση της Λιβύης. Σε αυτό το πλαίσιο το σώμα μας ξεκίνησε ε, μια εταιρική σχέση με τους ε, δημάρχους της Λιβύης που είναι η μόνη δημοκρατικά εκλεγμένη αρχή να δημιουργήσουμε δυνατότητες και να βρούμε λοιπόν νέους εταίρους αυτή είναι η προσπάθειά μας τα δικά μας μέλη δήμαρχοι από τη Φλάνδρα και τη Μούρθια από το Μέχελεν, την Τριέστε, τη Βιαρέλ και την Λευκοσία καθώς και πολλοί άλλοι βοηθούν σήμερα τους Λίβιους συναδέλφους τους οργανώνουν ασκήσεις, ε, προγράμματα κατάρτισης για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στην Λιβύη. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι όταν μιλάμε για τη διαχείριση της μετανάστευσης πρέπει να έχουμε κατά νου για το θέμα της ένταξης. Οι τοπικές δράσεις παντού στην Ευρώπη χρειάζονται. Πολύ σημαντική επίσης η ανθρωπιστική δράση και πολλοί από τους εθελοντές μας ε, συνεργάζονται με αυτές τις δράσεις. Βεβαίως πρέπει να βρίσκονται λύσεις οι οποίες να ταιριάζουν με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, με τις τοπικές παραδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και πολλοί πολίτες οι οποίοι εθελοντικά ε, βοηθούν, προσπαθούν να συνδράμουν τους, ε, τις αρμόδιες αρχές. Θέλω να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά τον πρόεδρο Ταγιάννη που πήρε την πρωτοβουλία αυτή Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μάρκουλα γιατί υποστηρίξατε την ε, εργασία των ε, τοπικών αρχών, των περιφερειών, νομαρχιών και ούτω καθεξής για την επίλυση της αποδοχής ε, προσφύγων και μεταναστών. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, ο κύριος Ντάσης γιατί μιλάμε και για την κοινωνική διάσταση του ζήτηματος. Όπως ε, είπαν και οι προλαλήσαντες. Ας ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε Ταγιάννη. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία σας διοργάνωσης αυτής της μεγάλης ε, διάσκεψης για το θέμα της ε, μετανάστευσης που απασχολεί όλες μας τις κοινωνίες. Ευχαριστώ που καλέσατε και την ΕΟΚΕ να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διάσκεψη. Είναι και πολλοί συνάδελφοί μου στην αίθουσα. Το θέμα αυτό είναι πανταχού παρών και επηρεάζει την πολιτική ζωή όλων των χωρών. Η ΕΟΚΕ εδώ και πολύ καιρό έχει ταχθεί υπέρ μιας νέας νόμιμης μεταναστευτικής πολιτικής και ενός αποτελεσματικού προγράμματος χορήγησης ασύλου που να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Θα πρέπει όμως να γίνει διάκριση μεταξύ των προβλημάτων των ε, προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Ως προς τους πρόσφυγες, εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι, γιατί μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για τον χώρο ελευθερίας και τα θεμελιώδη μας δικαιώματα. Θα πρέπει να χορηγήσουμε άσυλο σε ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο και το θάνατο. Επίσης και από νομικής πλευράς είμαστε υπεύθυνοι γιατί όλοι έχουμε συνυπογράψει την Σύμβαση της Γενέβης το 1951. Αυτή η σύμβαση τότε είχε υπογραφεί για να υποδεχτούμε τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και μερικές από αυτές τις χώρες τώρα αρνούνται να υποδεχτούν ε, μετανάστες. Μιλάμε ε, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πλέον και με βάση την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ε, επανεγκατάστασης 160.000 μεταναστών αφορούσε την ένταξή τους που αποτελεί το 0,035% του συνολικού πληθυσμού. Είναι κρίμα που δεν γίνεται η επανένταξή τους γιατί αλλού ε, είναι χώρες ε, υπεύθυνε να υποδεχτούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, διότι έχουν κινήσει τη διαδικασία ε, επί παραβάση κατά των χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης αυτών των μεταναστών. Θα πρέπει να γίνει μία αποτελεσματική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και να εκινήσουμε με μια κοινή διαδικασία με εγγυήσεις που να είναι ε, αξιόπιστες και ευέλικτες έτσι ώστε να υπάρχει νόμιμη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ανθρώπων που είναι θύματα διώξεων. Σε σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχουν ε, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που θα ήθελαν να μεταναστεύσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην είμαστε υποκριτές. Δεν μπορούμε να υποδεχθούμε όλα αυτά τα ε, εκατομμύρια με βάση τη δημοκρατική μας κατάσταση. Χρειαζόμαστε μετανάστες, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί μία ρύθμιση της μετανάστευσης. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία με τρίτες χώρες. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η συνεργασία, και για να καταπολεμήσουμε τις ρίζες της ε, ε, κακοδαιμονίας, πέρα από τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής και η ύπατη εκπρόσωπος. Πέρα από αυτές τις επενδύσεις λοιπόν που είναι απόλυτα αναγκαίες σε αυτές τις χώρες, δεν πρέπει να αγνοούμε και την πολιτική και θεσμική καθώς και διοικητική διάσταση του ζητήματος της σταθερότητας και ευημερίας σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε αυτή την στρατηγική για την επίλυση των σειράξεων και την ενδυνάμωση των κρατών, την πρόθεση της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές. Σε σχέση τώρα με την εποπτεία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει τα περιφερειακά κράτη του Νότου κυρίως, αύριο μπορεί να είναι οι χώρες του Βορρά ή της Ανατολής, της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν θα πρέπει να φέρουν λοιπόν αυτές οι χώρες μόνο την ευθύνη περιφρούρησης των συνόρων. Η ΕΟΚΕ χαιρέτησε την ενίσχυση της Frontex, αλλά θα πρέπει να επιτελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος σε αυτό το τομέα, πρόοδος που σχετίζεται και με μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Σε σχέση με την υποδοχή και ένταξη προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει να προωθήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων και η ένταξή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής κοινωνικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες και θα πρέπει να μπούμε στη θέση τους. Για παράδειγμα, ε, να δούμε τι γίνεται με ένα συνταξιούχο που έχει μία πολύ χαμηλή σύνταξη ή με μία ανήπαντρη μητέρα που έχει παιδιά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς εντάσσονται και αυτοί οι πρόσφυγες σε σχέση και με πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και μιζέριας. Θα πρέπει λοιπόν να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τους μετανάστες. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ανθρωπιστικό θέμα των μεταναστών από την απαρχή της κρίσης. Γιατί, γι' αυτό και το Δεκέμβριο του 15 και Ιανουάριο του 2016 μεταβήκαμε σε 11 κράτη-μέλη για να έρθουμε σε επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να δούμε ποιες είναι οι επιτυχίες ή αποτυχίες και οι χρηστές πρακτικές αυτών των φορέων στην ε, κρίση, στο προσφυγικό. Επίσης, θα πρέπει να καταρτήσουμε ευρωπαϊκές ε, πολιτικές. Δεν ε, είμαστε κάτοχοι της αλήθειας, αλλά θα πρέπει να προωθούμε ένα μόνιμο διάλογο με όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η πρότασή μας θα πρέπει να είναι σύνθεση όλων των απόψεων. Θα πρέπει να βρούμε συνετές λύσεις και όσοι λαμβάνουν αποφάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτά τα δεδομένα και να είναι γνώμονάς τους. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Πρόεδρε. Και πριν λήξει αυτός ο πρώτος κύκλος, ο κύριος Τούρκα έχει το λόγο εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών και των, ε, της, ε, του Οργανισμού για, τους, ε, για την ύπατη των ύπατων προσφύγων. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Είναι η ευκαιρία λοιπόν για μας να γιορτάσουμε τη ε, έκδοση των αιτήσεων στατιστικών στοιχείων και αυτό μας επιθυμίζει ότι όντως ο κόσμος βρίσκεται σε α, κρίση. 65,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι λόγω σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκρούσεων και βία. Είναι σημαντικό όμως να αναλύσουμε και τα στοιχεία αυτά. Δύο τρίτα των 65 εκατομμυρίων είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, πάνω από 40 εκατομμύρια. Δεν μπορούν να φύγουν καν από τη χώρα τους. Από τα 17 δισεκατομμύρια άμα, πρόσφυγες που απασχολούν την υπηρεσία του ΟΗΕ, 84% ζουν στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου και δεν καταφτάνουν στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας δώσω τρεις σκέψεις μαζί σας, ε, πολύ σημαντικές πιστεύω. Καταρχάς, ε, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας είναι το άσυλο, η προστασία σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Η σύμβαση του 51 που κατοχυρώνει αυτή την παράδοση. Να μην ξεχάσουμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο κατασκευάστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ευρώπη μάλιστα. Κατά δεύτερον, οι πρόσφυγες μας επενθυμίζουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου αλληλεξαρτέμαστε όλοι, όπου το τοπικό επίπεδο συναντιέται με το παγκόσμιο και έχουμε εδώ πολλούς δημάρχους, πολλούς επιτρόπους που εργάζονται καθημερινά στο πιο ε, τοπικό επίπεδο για να κάνουν ε, τα όσα χρειάζονται για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κάποιοι αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες ως μία απειλή για την ταυτότητά τους. Κάποιοι από αυτούς που αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες ως απειλή δεν τους έχουν γνωρίσει ενδεχομένω ποτέ. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να τους ε, ε, κάνουμε να καταλάβουν ότι οι πρόσφυγες δεν είναι άνθρωποι που να πάρουν, έρχονται να πάρουν κάτι. Μπορούν να συμβάλλουν. Μπορούν να συμβάλλουν αν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και αν υπάρχουν σωστά προγράμματα για την ενσωματώσή τους. Δεν είναι λοιπόν ε, δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 46 ήδη α, ανακήρυξε το θέμα των προσφύγων ως θέμα α, διεθνούς σημασίας και τρίτον και πρόκειται για την τελευταία σκέψη που θα σας παρουσιάσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο μοναδικός δρόμος για το μέλλον είναι η πολυμέρεια. Είναι προς το συμφέρον όλων των εθνικών κυβερνήσεων να συνεργαστούμε σε ένα πολυμερές πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκατε και δείξατε και στον υπόλοιπο κόσμο το πώς γίνεται αυτό και μάθαμε το 2015 τα διδάγματα. Παρουσιάσαμε μία σειρά προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κρατημέλη σε ό,τι αφορά το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την εξωτερική δραστηριοποίηση. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας επ' αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανέφερε η κυρία Εμπορ πρόκειται για μία μοναδική πραγματικά ευκαιρία για να δοθεί πνοή σε αυτό που εγκρίθηκε πέρσι στη Νέα Υόρκη, στην Σύνοδο των Ηγετών με την διακήρυξη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η Γενική Συνέλευση μας ζητά να αναπτύξουμε παγκόσμια αρμοδιότητα για τους πρόσφυγες και πραγματικά πρέπει να το πετύχουμε αυτό και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για το πώς θα τα πετύχουμε αυτά γιατί πραγματικά από αυτό εξαρτάται και το μέλλον της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your contribution. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας, κύριε Τουρκ. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕ, ο κύριος Καναπιακό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε του Κοινοβουλίου πρόεδρε της Επιτροπής, εξοχότητες. Όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσπαθεί να παίξει το ρόλο της ενισχύοντας την εξέβρεση λύσεων στο πρόβλημα της μετανάστευσης, προσπαθούμε να δράσουμε εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που αποσχολεί συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μακροοικονομική ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμα ώστε οι χώρες που αντιμετωπίζουν την οικονομική αστάθεια να γνωρίσουν περισσότερη ανάπτυξη και μόνιμη τάση προς την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί ε, ε, σκληρά με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα ε, για να αντιμετωπίσουμε σε ειδικέ περιστάσει όσα συμβαίνουν. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την πείρα μα γιατί είμαστε ο μεγαλύτερο πολυμερή οργανισμό και εντό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε δράση για να καλύψουμε τι ανάγκε μα. Το 2016 οι επενδύσει μα φτάσαν τα 84 δι, εκ των οποίων 8,4 αφορούσαν έργα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και των συνόρων τη. Η ΕΤΕ στήριξε τον τελευταίο χρόνο δράση εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιε από αυτέ είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ασφαλέστερο πόσιμο νερό και καλύτερο σύστημα απευθύνση σε 6,2 εκατομμύρια ανθρώπου με χιλιόμετρα ε, ασφαλών δικτύων 300.000 νοικοκυριά να διασυνδέονται με βιώσιμα μέσα και επίσης χιλιάδες επιβάτες να έχουν ασφαλέστερες μεταφορές. Όλα αυτά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω. Αυτές οι επενδύσεις ε, στα πλαίσια της οικονομικής ε, αντοχής μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα τα γενεσιογράτια της μετανάστευσης. Όμως πρέπει και θα δώσουμε και περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αρχή τις προσπάθειες των εθνικών και τοπικών αρχών να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές ροές με ιδιαίτερες ευθύνες ε, να αναλαμβάνονται από τα κράτη-μέλη για επενδύσεις σε σχέση με τους μετανάστες. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στηρίζουμε το Βραδεμβούργο, το γερμανικό αυτοκρατήδιο, για να χτίσει υποδομές που θα γίνουν αργότερα στέγαση, σημείο που θα μπορούν να υποδεχτούν συγκεκριμένε ομάδες πληθυσμού. Στα νότια Βαλκάνια, ε, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προχωρήσαμε την πρωτοβουλία για την οικονομική εντοχή και ανθεκτικότητα. Η πρωτοβουλία αυτή θα σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη από την ΕΤΕ στις δύο ενδιαφερόμενες περιοχές. Πέραν του δικού μας, ε, της δικής μας τακτικής δανειοδότησης, η διευκόλυνση προβλέπει πλέον 6 δι χρηματοδότηση για σκοπού οικονομική ανθεκτικότητας, ελπίζοντα ότι θα έχουμε 50 δι ευρώ περισσότερε επενδύσει ω το 2020. Η κινητοποίηση των επενδύσεων θα φτάσει τα 35 δι, ελπίζουμε. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να υπάρξει το πρώτο βήμα του πρώτου σκέλου για την ε, ε, προσπάθεια αύξηση των επενδύσεων βάσει του επενδυτικού προγράμματο. Τα βήματα αυτά προόδου συνοδεύονται από νόμου για τι μικρομεσαίε με 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ιορδανία, την Αιγύπτο, το Λίβανο, το Μαρόκο και την ε, Δυτική Οχθή. Και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν 38.000 θέσει εργασία στην Αφρική. Μαζί με την πρεσβεία του ΟΗΕ έχουμε το σχετικό πακέτο μέτρων για τη μετανάστευση με μέτρα υψηλότερου επίπεδου για να βοηθήσουμε τι φτωχότερε κοινότητε να προχωρήσουν γρηγορότερα με κοινοτόμε επενδύσει όπω την οικοδόμηση ουρανοξυστών που να ε, ε, ζεσταίνονται να καλύπτουν τι ανάγκε του ενέργεια από την ηλικιακή ενέργεια αλλά και την πρόσβαση των φτωχότερων κοινοτήτων τη υπαίθρου σε πόρου. Ε, εδώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιεργά αίτια τη μετανάστευση. Η επιτυχή διαχείριση τη μετανάστευση σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα, οι τοπικέ αρχέ και φορεί και οι χώρε εταίροι αλλά και τα ε, χρηματοοικονομικά ιδρύματα παγκοσμίω καθώ και η παγκόσμια κοινότητα θα συνεργαστούν με τρόπο αποτελεσματικό. Αναμένουμε αυτή τη συνεργασία και να μην ξεχνάμε ότι η ΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη πολυμερή τράπεζα που δράσει στην περιοχή. Έχουμε επαφέ ε, επιτόπου στην πράξη και γνωρίζουμε τα έργα που αναπτύσσονται. Ξέρουμε τι γίνεται με τους νόμους ε, και τις δωρεές μας και μπορούμε να προσφέρουμε τεχνική στήριξη που τόσο πολύ χρειάζεται στη φάση προετοιμασίας των προγραμμάτων και την εκτέλεσή τους. Έχουμε την ε, τεχνογνωσία για να μπορέσουν όλα αυτά να λάβουν σαρκα και Με τη δική σας τη συνεργασία και την εταιρική μας σχέση ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο στους ανθρώπους αυτών των περιοχών για να οδεύσουμε προς την ευημερία και να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος όπως είπατε και εσείς κύριε Ταγιάννη. Πάνω απ' θέλω να τους δώσουμε ελπίδα. Ευχαριστώ. Grazie mille, ringrazio tutti Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ε, έγκριτους προσκεκλημένους μας που ε, συμμετείχαν σε αυτή την ανακτήρια φάση της ε, ημέρας αυτής, της ημερίδας για τη μετανάστευση. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και όλους τους υπαλλήλους του Ευρωκοινοβουλίου που συνέβαλαν στην διοργάνωση αυτής της ημέρας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ευχαριστώ και τους συνεργάτες ε, του γραφείου μου και όλους όσοι ενεργά έλαβαν μέρος για να γίνει αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Τώρα θα περάσουμε στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου Γιούνκερ, τη είπατε εκπροσώπου Μογκερίνη και μου το ιδίω στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου. Ταυτόχρονα ξεκινούν αμέσω οι συζητήσει του Αγγελή Τράπεζα. Πρώτα απ' όλα διαχείριση του άσυλου και τη μετανάστευση σε αυτήν την αίθουσα, όπου θα προεδρεύσει ο Πρόεδρο ε, τη Επι... Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων, ο κ. Ε, Μωράη ενώ η άλλη θα γίνει στην ακριβώς απέναντι αίθουσα, την αίθουσα 3 50, στην οποία θα προεδρεύσει η πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, η κυρία Μακάβα. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Μωράης για να περάσουμε σε αυτή τη φάση της συζήτησης. ευχαριστώ.